ε, ξεκινήσουμε τη σημερινή ε, συνεδρία ψηφοφοριών. Καταρχάς πρέπει να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Ε, ο πρόεδρος έλαβε από τους σοσιαλιστές ε, καθώς και από τη γραμματεία των μη εγγεγραμμένων προτάσεις για ορισμούς, δύο ορισμούς που πρέπει να σας αναγνώσω. Για την Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και ενέργεια, ο κ. Μασιμιριάνο Σαλίνη στη θέση του κ. Αντώνιο Ταγιάννη. Ε, αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Βραζιλία η κυρία Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη στη θέση του Κύριο Αντώνιο Ταγιάννη. Είναι αντιπροσωπεία με το Περκόσουρ, ο κύριος Σαλβατόρ Ντομένικο. Για την αντιπροσωπεία. Λατινοαμερικής ο κύριος Σαλβατόρης, θέση του κυρίου Αντώνιο Ταγιάννη. Για την Ένωση του Αραβικού Μαγρέτ η κυρία Αγιάλα Σέντα στη θέση της κυρίας Έλενα Βαλεντιάνο για την ε, αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής η κυρία Νέσα Γελασάντερ, Σάντερ στην κυρία θέση της κυρίας Βαλενσιάνο για την ε, συνέλευση της ε, Ευρωμεσογειακής η κυρία Σέντερ για την κυρία Βαλενσιάνο για την αντιπροσωπεία Euronest την κυρία Γραπίνη και τέλος για την Επιτροπή των Αναφορών η κυρία Ντάιαν Τζέιμς, στη θέση του κυρίου Ζαν Μαρί Λεπέν Παρατηρήσεις? Όχι δεν υπάρχουν. Οπότε εγκρίνονται ε, αυτοί οι διορισμοί.